Καλό απόγευμα αγαπητοί συνάδελφοι. Αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα πρώτα να δώσω το λόγο στον κύριο Μάρκο Σέλο που είναι ο επικεφαλής αντιπροσωπείας με το, το Ισραήλ.